να προαχθεί και όχι να περιστεί το έργο των ε, ενεργών ΜΚΟ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη είναι η προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή κατάσταση στον Ιορδάνη ποταμό με ειδική αναφορά στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη ποταμού. Ο συντάκτης της ερώτησης, ο κύριος Δεκάστρο, έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο ποταμός Ιορδάνης εκπροσωπεί ένα μεγάλο ε, μέρος της κληρονομιάς μας, όχι μόνο περιοπλοντικής άποψης, αλλά και οικονομικής ε, για τα Παλαιστινιακά εδάφη, την Ορδανία και το Ισραήλ. Η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί παρά να μα ανησυχεί. Διότι πρέπει να επισημάνουμε ότι περίπου 98% του 1,3 δεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικών γλυκών υδάτων του ποταμού ε, εκτρέπεται ετησίω. Και υπάρχει και κίνδυνο αποστράγγιση. Εδώ λοιπόν μιλάμε για κινδύνου προ τη βιοπικιλότητα καθώ και πρόσβαση των τοπικών πληθυσμών στι πηγέ νερού διεθνεί διαπραγματευτές καθώς και η Αμερικανική, το Αμερικανικό Κοινοβούλιο, η Ευρωμεσογειακή Εθνοσυνέλευση ζήτησαν παρέμβαση. Παρέμβαση όχι μόνο των κυβερνήσεων και των τοπικών αρχών των τριών αυτών χωρών αλλά και του Συμβουλίου της Επιτροπής και των Κρατών Μελών ώστε να δοθεί τεχνική και οικονομική βοήθεια για την εξυγίανση του ποταμού. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στο κοινό ψήφισμα που προσυπογράφουν όλες οι πολιτικές ομάδες και τι οποίε ευχαριστώ για τη στήριξή του. Ζητούμε από την Επιτροπή να προβλέψει ένα σαφές και ακριβές, μια ακριβή και σαφή αναφορά στο σχέδιο αυτό και στα πλαίσια της πολιτικής γυπνίασης ε, με το Ισραήλ και τις Παλαιστινιακές, την Παλαιστινιακή Αρχή. Ένα πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι η κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων του Ιορδάνη ποταμού. Γνωρίζουμε ότι τα νερά είναι, το νερό είναι ένα αγαθό πολύτιμο για όλη την ανθρωπότητα και θέλω να επισημάνω την προσοχή σα ότι η ορθή κατανομή στο γεγονό ότι η ορθή κατανομή του νερού ε, για τη δίκαιη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού είναι ένα δικαίωμα που δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε. Είναι ένα θέμα λοιπόν ύψη τη σημασία για να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Α ε, ατενίσουμε λοιπόν με ελπίδα τι ειρηνευτικέ διαπραγματεύσει που ξεκίνησαν μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνη πρόσφατα και α ε, δούμε πώ μπορούμε να διαχειριστούμε του υδρολογικού πόρου κατά τρόπο ε, αποτελεσματικό. Έτσι, ώστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να οδηγηθούμε σε αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, των τοπικών κοινοτήτων και των οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών στι χώρε και τα εδάφη που, που ενδιαφέρονται για την λεκάνη του Ιορδάνη και βρίσκονται γύρω από τη λεκάνη του Ιορδάνη ποταμού όχι μόνο για το μέλλον του ίδιου αυτού του ποταμού, αλλά και για να με βελτιώσουμε τι συνθήκε διαβίωση των τοπικών πληθυσμών. Σα ευχαριστώ. Εξ ονόματο τη Επιτροπή, ο Επίτροπο ο κ. Φιούλε για λεπτά. Oh, Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μας δώσατε σήμερα να συζητήσουμε για το θέμα του Ιρδάνη ποταμού. Όντως, το θέμα των υδάτων στην περιοχή είναι πηγή ανησυχιών. Και ακούω και τις ανησυχίες των ευρωβουλευτών εδώ εξαιτία των προβλημάτων που υπάρχουν έλλειψης ύδατος στην περιοχή ή εξαιτία της κακής ποιότητας των υδάτων. Γνωρίζουμε τι συνέπειες μπορεί να έχει κάτι τέτοιο και περιβαλλοντικές ε, αλλά και ασφάλειας στην περιοχή. Πιστεύουμε ότι αποτελεί προτεραιότητα το νερό για την περιοχή. Είναι μια μεγάλη πρόκληση που απαιτεί λύση. Επίσης γνωρίζουμε πολύ καλά και γνωρίζετε κι εσείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φροντίσει να αναλάβει βήματα υπέρ των ειρνευτικών συζητήσεων μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Το νερό είναι ένα από τα θέματα που θα κληθούν να λύσουν οι δύο πλευρές πέρα από την Ιερουσαλήμ την ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι είναι ιδιαίτερη κατάσταση όσον αφορά τον κάτω Ιορδάνη και ξέρει ότι χρειάζεται καλύτερη διαχείριση των υδάτων εκεί από όλες τις πλευρές και των πηγών επίσης του Ιορδάνη. Γι' αυτό και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο έχουμε αναλάβει δραστηριότητες με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Στηρίζουμε μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που θα βοηθήσουν να υπάρχει βιωσιμότητα στην περιοχή όσον αφορά το είδωρ. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης γυτνίασης αλλά και άλλα μέτρα θέλουν να υπάρξει οικοδόμηση εμπιστοσύνης με διασυνοριακή συνεργασία και φέρνοντας τις πηγές του ύδατος να τυχαίνουν διαχείριση από όλε τι πλευρέ. Οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως στόχο την οικοδόμηση ικανοτήτων από όλε τι πλευρέ που διαχειρίζονται το είδωρο στην περιοχή όπως επίσης είναι υπέρ και της συλλογής στοιχείων, ε, επεξεργασίας ε, λιμάτων, αλλά και μέτρων ε, προστασίας του ύδατος. Επίσης είμαστε και υπέρ μέτρων που θα βεθίσουν την σωστή άδρευση στην περιοχή. Θέλουμε να υπάρξουν συνθήκες εκείνες οι οποίες θα επιτρέψουν μια ολοκληρωμένη διαχείριση των πηγών ύδατος στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι βέβαια μόνη τη σε αυτή τη δουλειά και σε αυτή την προσπάθεια και άλλες χώρες και άλλοι δωρητέ βοηθούν. Συντονίζουμε λοιπόν τις δραστηριότητές μας μαζί τους προκειμένου να διασφαλίσουμε συμπληρωματικότητα στις δράσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Εξ των πολιτικών ομάδων, πρώτα η κυρία Κράτσα για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε κύριε επίτροπε κύριε και κύριοι συνάδελφοι είναι πολύ θετικό βήμα ότι αναδεικνύεται η πρόκληση του ιορδάνη ποταμού σήμερα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. η ευρωμεσογειακή κοινοβουλευτική συνέλευση έχει εκπονήσει ειδική μελέτη για τα θέματα του ιορδάνη και της κοιλάδας του και έχει κάνει έκκληση για την προστασία του στα ψηφίσματά της γιατί ο ιορδάνης ποταμός είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς αποτελεί σύμβολο θρησκευτικό πολιτισμικό για εκατομμύρια πολίτες στον κόσμο και ένα κεφάλαιο οικολογικό τουριστικό οικονομικό ε, για τους κατοίκους της περιοχής. στόχος λοιπόν σήμερα είναι να αναδειχθούν τα προβλήματά του και η ανάγκη κινητοποίησης για την προστασία του εντατικοποίηση των προσπαθειών που κάνει η ευρωπαϊκή ένωση, ένωση αναφέρθηκε σε αυτά ο επίτροπος τα έχουμε θίξει και με άλλες ευκαιρίες σε συνεργασία με την κοινή γνώμη ε, να γίνει μια έκκληση για την ε, περιφερειακή συνεργασία για τη δίκαιη πρόσβαση των λαών που βρέχονται, λαών που βρέχονται από τον Ιορδάνη και ε, τον καταμερισμό ευθυνών για την προστασία του. Το ψήφισμα που προτείνεται αναδεικνύει και καλές πρακτικές όπως το ένα master plan ειδικό που έχει εκπονήσει ε, ε, το Ισραήλ και ζητείται η ανταλλαγή καλών πρακτικών η ανταλλαγή τεχνογνωσίας διότι αποτελεί μια συλλογική υπόθεση της περιοχής επίσης ε, είναι σημαντικό ότι αναδεικνύονται ε, οι, πραγματικοί κίνδυνοι που δεν είναι μόνο η στέρηση των υδάτων δεν είναι μόνο η μόλυνση αλλά είναι η απώλεια της βιοποικιλότητας ο κίνδυνος της αποξήρασης μάλιστα αν συνεχίσουμε την ίδια κατάσταση. και για να ε, αναδειχθεί αυτή η διεθνή συνεργασία η περιφερειακή συνεργασία στο ψήφισμα προτείνεται και μια ειδική επιτροπή για την κοιλάδα του ιορδάνη ε, στην οποία ε, ε, θα, έχουν, μπορούν να λάβουν μέρος οι χώρες, που άμεσα έχουν σχέση με τον Ιορδάνη, Ισραήλ, Παλαιστινιακά εδάφη, Ιορδανία, αλλά και άλλες χώρες της περιοχής, εκεί που ε, ξεκινάει ο ιορδάνης και που έχουν και αυτές μερίδιο ευθύνης όπως είναι ο λίβανος και η συρία. πιστεύω ότι θα τύχει υποστήριξη της ε, ολομέλειας στο ψήφισμα αυτό και θα είναι μια ε, συγκροτημένη στοχευμένη και δυνατή φωνή αυτή που θα στείλει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ακούσαμε, η κατάσταση της νεκράς θάλασσας και του ποταμού Ιορδάν είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Προβλέπετε ότι αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, πολύ σύντομα μπορεί να στερέψει τελείω ο ποταμός. Έτσι λοιπόν, είτε σε διεθνές είτε σε περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να αναλάβουμε δράση για να σταματήσουμε αυτή την πορεία να την ανακόψουμε προκειμένου να μην έχουμε απώλεια, ε, μια απώλεια εξαιρετικά σημαντική και για τη γεωργία και για τη βιοπικιλότητα, όπως είπε η κυρία Κράτσα. Και για την ασφάλεια της οικονομίας και την οικονομία της όλης περιοχής. Εδώ να θυμίσω μια με κυβερνητική οργάνωση που ανέλαβε μια εξαιρετική, κατά την άποψή μου, πρωτοβουλία. Η οργάνωση Friends of the Earth στην Μέση Ανατολή και η οποία αποφάσισε να συγκεντρώσει τους δημάρχους της ε, Παλαιστίνης, της Ιορδανίας και του Ισραήλ που βρίσκονται στις όχθες του, των, των κέντρων, αστικών κέντρων που βρίσκονται στις όχθες του ποτάμου. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν για να συζητήσουν τι μπορούν να κάνουν για να βελτιώσουν κάπως τα πράγματα. Και σε αυτή τη συνάντηση, μαζί με τους δημάρχους, επώνυσαν μελέτες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Δηλαδή, τι μπορεί να συμβάλλει κάθε χώρα στη λύση του προβλήματος, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος των μέτρων που θα αναλυθούν και τι θα μπορούσε να γίνει μέχρι και η αλλαγή των γεωργικών μεθόδων, το είδος των καλλιεργιών που απορροφούν πολύ μεγάλο ποσό νερού και ούτω καθεξής. Να τι μπορεί να κάνουν λοιπόν κάποιες φορές και οι πολίτες. Εδώ η συζήτηση αυτή έχει και πολιτικό βέβαια χαρακτήρα αλλά όχι ακρεφνώς, παρόλο που όποτε μιλάμε για νερό στην περιοχή αυτή, εννοείται ότι υπάρχει και πολιτική φύση στο πρόβλημα. Πρέπει να πω πάντως σε κάθε περίπτωση ότι η Ευρώπη και η Επιτροπή πρέπει να εμπνευστούν από τα πολύ σαφή συμπεράσματα της έκθεσης αυτής και στις σχέσεις τους με τις τρεις παραποτάμιες χώρες. Πάντω υπάρχει και ένα συγκεκριμένο εδάφιο, το ε, το οποίο μου είναι ιδιαίτερα προσφυλέ, διότι λέει ότι υπάρχει υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων από του Ισραηλινού επίκου. Αληθεύει αυτό και το αποδεικνύει και η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Amnesty International είναι και θέμα της Διεθνούς Αμνηστίας, είναι θέμα <clears throat> και πολιτικό και ίσως να μην είναι στο κέντρο του ψηφίσματός μας, αλλά είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. η για λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ως Αντιπρόεδρος της Ευρωμεσογειακής ε, για την ενέργεια των περιβάλλον και τα ύδατα, είχα την ευκαιρία να δω αυτή την τραγική πραγματικότητα στον Ιορδάνη κατά τη διάρκεια μια επίσκεψη που έλαβε χώρα πέρυσι το Φεβρουάριο, μάλλον αυτό το Φεβρουάριο. Ε, εγώ ήμουν εισηγήτρια για τον Ιορδάνη και διαπίστωσα ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, κυρίω ε, το Ισραήλ, η Παλαιστινιακή Αρχή και η Ιορδανία, αλλά και ο Λίβανο και η Συρία, όλοι πρέπει να βρουν μια λύση στο πιο πιστικό πρόβλημα που είναι η ίση κατανομή νερού, η οποία θα σέβεται τι ανάγκε όλων των ανθρώπων στην περιοχή ε, θα σέβεται το περιβάλλον που είναι σημαντικό για τις επόμενες γενιές. Ε, το πρώτο που βρήκα στην έκθεσή μας ε, και αναφέρεται είναι ότι οι Ισραηλοί και οι Παλαιστίνοι πρέπει να συμφωνήσουν για την τη ισομερή διαχείριση των υδάτων, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις γιατί και οι δύο πλευρές όπως και ανεξάρτητες εκθέσεις παρουσιάζουν διαφορετικά στοιχεία μέχρι τώρα. Ένα από τα βασικά μας συμπεράσματα είναι ότι για να λυθεί το πρόβλημα των υδάτων μέσα από τη συνεργασία είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα για την κοινή διαχείριση, τη λήψη αποφάσεων με ίσε προποθέσει, κοινή διαχείριση των υδάτινων πόρων στην περιοχή. Πιστεύω ότι η έκθεσή μα και οι συστάσεις ε, ταυτίζονται ε, με τομεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρα πολλέ ε, ειδικέ γνώσει και μπορεί να συμμετέχει ω παίκτη για να ανοίξει το δρόμο στο μέλλον. Και τελειώντα θέλω να σε επισημάνω ότι γίνονται προσπάθειε και για να ξεκινήσει μια συνολική συμφωνία ειρήνης όπου όλοι θα αναλάβουν ε, την ευθύνη να μην χρησιμοποιούν την κατάσταση στον Ιορδάνη για πολιτικούς και ιδεολογικούς ε, σκοπούς. Πιστεύω λοιπόν ότι η συζήτησή μας σήμερα θα εξυπηρετήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην περιοχή και θα οδηγήσει σε αμερόληπτα συμπεράσματα για την ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Η κυρία Άουκεν για 1,5 λεπτό, εκ μέρους των Πρασίνων. Øh, er Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με τις δύο προλαλήσασες. Ενώνω και εγώ τη φωνή μου για να πω ότι πολλοί ξεχνούν πώς έγινε δυνατόν να αναλάβουν και οι Παλαιστίνοι την ευθύνη. Πριν από το 1967, 50% της Λωρίδας της Γάζας από τότε ε, βρίσκεται υποκατοχή. 45% εξάλλου προβλέπονται από τετάφη για προστατευμένες ε, περιοχές. Το πρόβλημα με την κοιλάδα του Ιορδάνη είναι ακριβώς ότι δεν υπήρξε αντίδραση στις στρατιωτικές παρεμβάσεις που έγιναν. Και έχουμε ξεχάσει τα μέρη αυτά. Να λοιπόν το μάθημα που πρέπει να πάρουμε εμείς εδώ σήμερα. Οι Παλαιστίνοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάτι για να πιστήσουν την προσοχή του κόσμου απάνω τους. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν μπορεί να δράσει στην περιοχή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα έτσι όπως έχει η κατάσταση σήμερα. Πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν ε, το πρόβλημα αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους. Άρα πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση που να συμπεριλαμβάνει ε, στα πολιτικά θέματα όχι μόνο την Ιορδανία και το Ισραήλ, αλλά και τους Παλαιστινίους. Πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να δράσουν. Ο κύριος Τάνοκ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ε, το νερό είναι ένα φλέγον θέμα στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, οι αντιπροσωπείε από το Ισραήλ και την Παλαιστινική Αρχή αυτή τη στιγμή συζητάνε τα δικαιώματα στα ύδατα ε, στο πλαίσιο τη ε, Συμφωνία για την Ειρήνη η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να είναι εγγυητή στην περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην ε, επηρεάσουμε τι διαπραγματεύσει που τρέχουν αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον. Όπω είπε και αυτό που κάνει η κυρία Ντεκάιζερ, το να κατηγορούμε του Ισραηλινού επίκου για υπερβολική χρήση, κατάχρηση νερού, αυτό είναι ένα ε, μήνυμα που μπορεί να ερμηνευτεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προκατηλημένη. Πράγματι το θέμα είναι σημαντικό και δεν περιορίζεται μόνο ε, ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους. Οι εχθροί του Ισραήλ σε αυτή την αίθουσα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το θέμα αυτό στο πλαίσιο της εκστρατεία τους ε, για να υπονομεύσουν το εβραϊκό κράτος. Ε, βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να αντιμετωπίζεται από τους Ισραηλινούς ως ανάξια του ρόλου της που θα ήταν εταίρος στην ειρήνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρόβλημα δεν είναι ότι έχει μια άποψη η κυρία Ντεκάιζερ. Στην πραγματικότητα, το 1994 στη συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ιορδανία αποφασίστηκε να συνεργάζονται για να αποκατασταθεί ο Ιορδάνης και για να προστατευθούν οι περιβαλλοντικοί πόροι. Είναι και αυτή μια συμφωνία. Βέβαια θα μου πείτε μια παραπάνω συμφωνία που δεν τηρεί το Ισραήλ. Μα αυτό ακριβώ είναι το πρόβλημα που έχουμε με το Ισραήλ, ότι δεν τηρεί τι συμφωνίε που υπογράφει. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η πρωτοβουλία που ανελήφθη το 2008 από το ΣΥΡΑΚ, που έκανε έκκληση ε, για μια πρωτοβουλία υπέρ του Ιορδάνη, να πάρει μορφή. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να φτιάξουμε μια επιτροπή για την λεκάνη του Ιορδάνη ποταμού, που να περιλαμβάνει όλες τις παραποτάμιες χώρες που να δουλέψουν υπέρ της περιοχής, να προστατεύσουν περιβαλλοντικά την περιοχή και να δουλέψουν για μια λύση όσον αφορά το Ιδωρική. Οι Παλαιστίνοι για άλλη μια φορά έχουν αποκλειστεί από τη ζώνη ασφάλειας του Ισραήλ και της Ιορδανίας. Εντελώς δηλαδή από τον κάτω Ιορδάνη και την περιοχή εκεί την κατέχουν οι έπικοι. Και επειδή ακριβώς πρόκειται για κατοχή και με την κατοχή γίνεται και χρήση παράνομη των υδάτων εκεί, προστίθεται άλλο ένα πρόβλημα πέρα από το πολιτικό πρόβλημα που είναι οικολογικό. Το 2011 που θα αρχίσουν να λειτουργούν νέα κέντρα επεξεργασία ελλημάτων εκεί, ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει, να δώσει κίνητρα για να δημιουργηθεί αυτή η Επιτροπή για τη Λεκάνη του Ιορδάνη Ποταμού. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στου υπόλοιπου εγγραμμένου ομιλητέ. Πρώτα ο κύριο Πρέντα για δύο λεπτά. Uh, Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση για την κατάσταση uh, στον ποταμό Ιορδάν είναι πολύ σημαντική για τη δική μου την πολιτική ομάδα. Θα ήθελα λοιπόν uh, να προβάλλω και να χαιρετήσω ιδιαίτερα την παρέμβαση της συναδέλφου της κυρίας Κράτσα όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ε, επανειλημμένα έχουν επισημάνει την ε, επισφαλή κατάσταση στην ε, περιοχή του Ιορδάνη. Ο ποταμός αυτός μοιάζει να πνέει τα λίστια. Στις εφημερίδες των τύπων μπορεί κανείς να διαβάσει ότι παρά την κρίσιμη κατάσταση οι Ορθόδοξοι χριστιανοί εξακολουθούν να βαπτίζονται στα ύδατα του Ιορδάνη. Όμως ε, το 2011 ενδέχεται να μην υπάρχει πια νερό. Και αυτό θα είχε καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον και για τη νεκρή θάλασσα. Οι Παλαιστίνοι αλλά και οι Ισραηλοί θα υποστούν βέβαια τις συνέπειες. Θα αντιμετωπίσουν μια οικολογική καταστροφή. Οι συνάδελφοί μου επισήμαναν κάτι το οποίο χρήζει επιγόντως ε, λύσεις. Η κατάσταση του ποταμού Ιορδάνη έχει ιδιαίτερη σημασία για την συνεργασία στην περιοχή. Οφείλουμε λοιπόν να αποφύγουμε μια κατάσταση όπου μία και μόνο χώρα ε, θα ε, εκμεταλλεύεται το σύνολο των υδάτινων πόρων και θα ληστεύει τους ε, πόρους αυτούς από τις όμορες χώρες ο ποταμός Ιορδάνης μπορεί να γίνει σύμβολο συνεργασίας, οικονομικής αλλά και πολιτιστικής συνεργασίας. Αν βέβαια και εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση προς αυτή την κατεύθυνση. Τα υδάτινα αποθέματα ε, είναι ένα θέμα που ακόμα δεν έχει επιληθεί όσον αφορά την κατάσταση του Ιορδάνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να Προτείνω στον κύριο Τάνοκ να σκεφτείτε το εξή. Δεν είναι απλό να αγνοούμε την πραγματικότητα. Οι έπικοι γνωρίζουν πολύ καλά που εγκαθίστανται προκειμένου να έχουν καλή προμήθεια νερού. Και δεν είναι το μόνο πρόβλημα βεβαίως σε σχέση με το νερό στην περιοχή αλλά είναι μέρος του. Ο Ιορδάνης κάνει το 98% των υδάτων του, διότι υπάρχουν πολλές διαδικασίε και ενέργειες εκτροπής, μεταξύ των οποίων από το Ισραήλ. Τέσσερα κράτη, μεταξύ των οποίων και η Παλαιστινιακή Δυτική Όχθη, βρίσκονται στις όχθες του ποταμού. Είναι τα λεγόμενα παραποτάμια κράτη. Αν ο καθένας διαδραματίσει σωστά το ρόλο του στην περιοχή. Θα μπορούσε να γίνει ένας παράγοντας σταθεροποίησης ο Ιορδάνης, προκειμένου να έχουμε μια υγιή διαχείριση των υδάτων που είναι και θρησκευτικό και οικονομικό σπόρος για την περιοχή. Εσείς κύριε Τάνοκ φαίνεται να λέτε ότι οτιδήποτε, οτιδήποτε έχει να κάνει με επίκριση του Ισραήλ ισοδυναμεί με επίθεση κατά της χώρας αυτής. Όχι, η πραγματικότητα είναι διαφορετική κι άλλη έχουν ε, προχωρήσει σε εκτροπή των υδάτων του Ιορδάνη. Ε, ένα πρόσφατο σεμινάριο που οργάνωσαν οι σοσιαλδημοκράτες απέδειξε ότι κάποια στιγμή ο Ιορδάνης είχε 1,3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού που τώρα έχουν περιοριστεί σε 20, σε 20 εκατομμύρια ετησίως. Μιλάμε για ένα ποταμό σχεδόν νεκρό, εκτός και αν αναλάβουμε εμείς δράση. Η κυρία για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν ε, πολλές αιτιάσεις ε, και εδώ από το Κοινοβουλίο και εκτός του Κοινοβουλίου για το ότι εξετάζουμε το θέμα της ειρήνευσης σε λάθος χρονική στιγμή και η δική μου η κοινοβουλευτική ερώτηση κατατέθηκε όταν δεν γνωρίζαμε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις πρόκειτο να ξεκινήσουν. Ε, το θέμα το εξετάζω εγώ από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και το θέμα αυτό υπάρχει στο Κοινοβούλιο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι το κάτω τμήμα του Ιορδάνη να προστατευθεί από την πλήρη καταστροφή. Γι' σε αυτό το κάτω κομμάτι ο Ιορδάνης έχει γίνει όχι υποταμός αυλάκι είναι πια. Και όλοι οι επιστήμονες συμφωνούν ότι σε ένα ή δύο χρόνια αυτή η εκβολή του Ιορδάνη δεν θα υπάρχει πλέον. Εκείνο που με εκνευρίζει στο ψήφισμα είναι ότι η Παλαιστινική Αρχή, ε, όλοι αυτοί και η Ορδανία βρίσκονται στην ίδια ακριβώ ε, θέση. Αλλά εδώ μιλάμε για την ε, ζώνη σε τη γάμα ζώνη, όπου η Παλαιστινιακή Αρχή δεν έχει κανένα απολύτω δικαίωμα, ούτε και διοικητικό, ούτε και οποιοδήποτε άλλο. Η ε, Παλαιστινιακή Αρχή επιτόπου δεν μπορεί να κάνει απολύτω τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι σε άλλου πρέπει να απευθυνθούμε. Βεβαίω αναφέρθηκε ότι πρόκειται για ένα πολιτικό θέμα. Όταν μια χώρα και συγκεκριμένα το Ισραήλ ε, χρησιμοποιεί το 75% των υδάτων, ενώ το έχει πάρει ε, εντωμεταξύ από άλλε χώρε και κατ' ουσίαν δεν αφήνει πια καθόλου νερό στου Παλαιστινίου για να επιβιώσουν. Αυτό προφανώ και είναι πολιτικό θέμα. Δυστυχώ ε, υπάρχει κάποια συμφωνία, αλλά δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει συγκεκριμένα το πρόβλημα ότι οι Παλαιστίνοι προσπαθούν συνεχώ να κάνουν γεωτρήσει, οι οποίες καταστρέφονται από ε, τους Ισραηλινούς. Οι Ισραηλινοί δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα για τους Παλαιστινίους παρά μόνο για, τις παρα... για τους παράνομους επικισμούς. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ξεκινήσω τιμώντας την οικολογική οργάνωση που δεχτήκαμε στις Βρυξέλλες και όπου συμμετέχουν και Ζελενοί και Παλαιστίνοι και που μας παρουσίασαν πολύ καλά την κατάσταση στην περιοχή και ιδιαίτερα στον Ιορδάνη με τον κίνδυνο εξαφάνισή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μεγάλα ποσά σε προγράμματα ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή. Θα έπρεπε λοιπόν να ασχοληθεί περισσότερο με την εκπόνηση ενό σχεδίου υπέρ τη διάσωση του Ιορδάνου που θα συμμετέχουν όλε οι περιοχέ ε, εκεί. Η Ιορδανία, το Ισραήλ εκτρέπουν ένα μεγάλο μέρος του ποταμού, ενώ οι Παλαιστίνοι μόνο 5% των πόρων μπορούν να έχουν. Οι δε έπικοι από το Ισραήλ ξοδεύουν έξι φορές περισσότερο νερό από τους Παλαιστινίους, ιδιαίτερα για την εντατική γεωργία που ρηπαίνει επιπλέον και που έχει σαν στόχο να εξάγουν προϊόντα, γεωργικά προϊόντα προς την Ευρώπη. Η επέκταση δε των επικισμών αυτών πρέπει να πάψει. Όπως επίσης πρέπει να πάψει και η καταστροφή, όπως πριν από λίγες εβδομάδες φέτος το καλοκαίρι, ε, καταβλισμών που καταστρέφονται και χώροι και άνθρωποι. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ισότιμη κατανομή του ύδατος στην περιοχή και αυτό πρέπει να αποτελέσει δικιά μας προτεραιότητα. Ο κύριος ε, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επιτρόπε. Η περιβαλλοντική καταστροφή που σήμερα συζητούμε ξεπερνά το γεωγραφικό χώρο το συγκεκριμένο και αφορά όλη την Ευρώπη και εμά του Ευρωπαίους. Η βιώσιμη ανάπτυξη στην οποία πιστεύουμε είναι μια έννοια η οποία δεν μπορεί να υπόκειται μόνο σε διοικητικά μέτρα, αλλά χρειάζεται να σεβαστούμε και τι θρησκευτικέ πεπιθήσει και τα υπόλοιπα στοιχεία που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Οι πληθυσμοί και οι τοπικέ κοινότητε που πλήττονται από τα προβλήματα του Ιορδάνη, λόγω του χαμηλή στάθμη των υδάτων, είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Το να ε, σκεφτόμαστε παγκόσμια αλλά να δρούμε τοπικά είναι κάτι που το επαγορεύει η κοινή λογική. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει τοπική δράση ώστε να περιορίσουμε την υποβάθμιση της λεκάνης του Ιορδάνη και να μειώσουμε την αποστράγγιση των υδάτων. Το να δράσουμε είναι κάτι σημαντικό γι' αυτό και έχει αναλάβει νομοθετική και θεσμική δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η η προώθηση του θέματος στην Ευρωμεσογειακή Συνέλευση καθώς και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν και βεβαίως η αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου που ασχολείται με τις σχέσεις ε, των χωρών Μασρέκ θα πρέπει να προωθήσει την εξέταση των θεμάτων αυτών. Θα πρέπει λοιπόν η περιβαλλοντική άποψη να απασχολήσει τόσο τα παραποτάμιες χώρες αλλά όσο και να εμπλέξει τους τοπικούς πληθυσμούς στην επίλυση των προβλημάτων. Το ψήφισμα λοιπόν σωστά ζητά τη δημιουργία μια επιτροπή για τη διαχείριση την κοινή διαχείριση των προβλημάτων του Ιορδάνη, εκπροσωπώντα τι αρχέ και τα κράτη που διαχειρίζονται τα είδα του ποταμού αυτού. Και έτσι θα πρέπει ετησίω λόγου χάρη να, ε, εργα... να συναντήσει όπου η Επιτροπή αυτή να μοιράζεται τι εμπειρίε τη με τη διεθνή κοινότητα. Έπειτα η ανταλλαγή καλών πρακτικών σε ό,τι αφορά κοινοτικά κοινά προγράμματα με τη συμμετοχή Ιορδανών ε, και Παλαιστινίων και Ισραηλινών για ένα θέμα που αφορά ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και για την σωστή ε, για διαχείριση των υδάτινων πόρων, συγκεκριμένα της λεκάνης του Ιορδάνη. Και βεβαίως μια ευρύτερη προσπάθεια για την ειρηνική συνύπαρξη στην οποία θα μεταφραστεί και η διαχείριση των υδάτινων πόρων. Εδώ λοιπόν θα πρέπει άμεσα να αναλάβει η δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση στην όλη διαδικασία, να φροντίσει να υπάρξει μια ε, άμεση έναρξη νέου μορφή διαλόγου μεταξύ Παλαιστινική Αρχή και Ισραήλ, ώστε να λυθεί και το πρόβλημα αυτό ως μέρος του ευρύτερου διαλόγου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, το θέμα της αποξήρανσης του Ιορδάνη είναι ένα οικολογικό πρόβλημα το οποίο ε, επηρεάζει και θέτει σε κίνδυνο το σύνολο της ε, περιοχής. Ο ποταμός αυτός είναι ιδιαίτερα μολυσμένος, έχει πολλές ε, διαρροές και αυτό οδηγεί στο ότι αποδυναμώνεται σημαντικά η διαχείριση των υδάτων. Όπως είπαν και ορισμένοι από τους προλαλήσαντες, τα ύδατα σε πάνω από 95% χρησιμοποιούνται για ε, βιομηχανικούς και γεωργικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου η ροή των υδάτων έχει περιστεί σε λίγα κυβικά μέτρα το χρόνο. Χιλιάδες κυβικά προφανώς. Το νερό δεν είναι μόνο πηγή μιλοτσέρδος αλλά μπορεί να οδηγήσει και στη συνεργασία και στη δημιουργία εμπιστοσύνη στην περιοχή. Αυτό λοιπόν είναι κάτι σημαντικό ε, και αν μπορέσουμε τελικά να λύσουμε αυτό το πρόβλημα θα επιτύχουμε πάρα πολύ πιο πολλά από οτιδήποτε άλλο αν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα κάτω από άλλο πρίσμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η εξήρανση του Ιορδάνη που προχωράει σιγά σιγά είναι ένα από τα δράματα που αντιμετωπίζει η Παλαιστίνη σήμερα. Είναι πολιτικό το θέμα, μην το ξεχνάμε. Η Παγκόσμια Τράπεζα μας λέει ότι εδώ και δύο χρόνια 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι στη λωρίδα της Γάζας δεν έχουν πια χλώριο, που είναι αναγκαίο για να απολυμένεται το νερό. Ήδη πριν τους βομβαρδισμούς ε, υπήρχε αυτή η κατάσταση, φανταστείτε σήμερα τι γίνεται. Ο Ισραηλινός στρατός επιτίθεται στις εγκαταστάσεις, το νερό που φτάνει στους κατήχους δεν είναι κατάλληλο για κατανάλωση. Επίσης, 4 εκατομμύρια λίτρα νερό δεν περνάνε από καμία απολύμανση, χύνονται στην Μεσόγειο, επειδή ακριβώ έχουν καταστραφεί υποδομές ε, στην Γάζα. Η κυρία Στον πήγε στη Γάζα πολλές φορές, ναι. Αλλά πού είναι το πολιτικό της θάρρος να εφαρμόσει, να επιμείνει να εφαρμόσει το Ισραήλ τις απαιτήσει μας. Το Ίδωρ, όπως και η γη, δεν ανήκει μόνο στους Ισραηλινούς επίκους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να σταματήσει τη συμφωνία σύνδεσης με τη σημερινή Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία κοφεύει στα δικά μας τα αιτήματα όσο συνεχίζεται η κατοχή και οι επικισμοί που είναι παράνομοι. Όσο δεν υπάρχει δικαιοσύνη δεν θα υπάρξει ούτε ειρήνη. Κυρία Μπεναράμπατου, για ένα λεπτό δεν πρόσεξα τι είπατε. Και δεν πρόσεξα ότι ξεπεράσατε λίγο το χρόνο σας. Για ένα λεπτό τώρα η κυρία Μπένοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε από τη σημερινή συζήτηση ότι ο ποταμός Ιορδάνης έχει αξιοσημείωτη οικολογική, πολιτική και θρησκευτική σημασία. Είναι ένας ποταμός στρατηγικής σημασίας. Η χρήση του και η κατάχρησή του είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποδεχτούμε από το 1964 έχει αρχίσει εκτροπή των υδάτων όχι μόνο προς το Ισραήλ αλλά και από, τη, από το Λίβανο, τη Συρία, τον Ιορδάνη έχουν ξεκινήσει ανάλογες προσπάθειες. Πολλές χώρες λοιπόν με τις ενέργειές τους έχουν καταστρέψει τον ποταμό. Και το επισημαίνουν και όλοι οι οικολόγοι. Το οικοσύστημα έχει καταστραφεί πλήρω. Και μπορεί σε μερικέ δεκαετίε να μην υπάρχει τίποτε εκεί. Είναι γεγονός λοιπόν ότι το Ισραήλ και οι αραβικές χώρες της ε, περιοχής δεν έχουν καταφέρει να βρουν λύση. Δεν έχουν εξηγιάνει τον ποταμό. Είμαι πεπισμένη λοιπόν ότι πρέπει να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση και να πιέσει επιβάλλοντας λόγω χάρη κριτήρια για την ε, επιδότηση προγραμμάτων αναπτυξικής βοήθειας στην περιοχή, προκειμένου να ε, πιέσει για τη λύση των προβλημάτων του Ιορδάνη Ποταμού.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 Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ο ανταγωνισμός ε, για το νερό μπορεί να ε, οξύνει περισσότερο μία σύγκρουση στο Κασμίρ, παραδείγματος χάνει και εκεί έγινε το ίδιο ε, η διαμάχη ανάμεσα σε τοπικές φυλές. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ στον Κάτω Ιορδάνη. Κοιτάξτε Πρόεδρε, το να αυτός ο ποταμός θα μπορούσε να αυξήσει και τις προοπτικές ειρήνευσης. Ο ποταμός αυτός ε, έχει ιδιαίτερη ιερή σημασία για τους ε, χριστιανούς αλλά και για τους ε, μουσουλμάνους οι Ισραηλοί έχουν διασχίσει τον Ιορδάνη και εκεί έγινε το θαύμα όπου ο Χριστός ε, περπάτησε πάνω στα νερά και δεν πρέπει να ε, να εμποδίζουμε να λάβει σήμερα ένα άλλο θαύμα, να λάβει χώρα ένα άλλο θαύμα, να ζουν οι άνθρωποι εν ειρήνη και αρμονία στην περιοχή. Ε, την κυρία Μπασέσκου, τον κύριο Μέντσιου και τον κύριο Μόλτσερ. Υπάρχει κάποιο άλλο. No one else. Very well. Ms. Basescu, one minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Consider că o rezoluție, o abordare părtinitoare a situației râului Νομίζω ότι ένα ψήφισμα το οποίο θα είναι κομματικό και θα τοποθετείτε για το θέμα του Ιορδάνη ένα τέτοιο ψήφισμα ε, δεν θα βοηθούσε στην υπόθεση της ειρήνης. Είναι ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο και κάποια στιγμή το πρόβλημα του κάτω Ιορδάνη πρέπει να διαλευκανθεί αλλά όχι τώρα που τρέχουν διαπραγματεύσει ειρήνευσης. Πρέπει λοιπόν να συναυθεί μια περιφερειακή συμφωνία στην ε, περιοχή. Εμείς ε, θεωρούμε ότι η περιφερειακή συνεργασία είναι καθοριστική σημασίας. Όλες οι παρόχθιες ε, χώρες πρέπει να συνεργαστούν. Τα 61 από τα 96 προγράμματα που εφαρμόζονται στην περιοχή δεν αφορούν τον Ιορδάνη, αφορούν γενικότερα θέματα και όχι τη ροή του Ιορδάνη. Το πρόβλημα της αποκατάστασης ε, του Ιορδάνη έχει πάρα πολλές ε, διαστάσεις. Ε, ο ποταμός Ιορδάνης έχει ιστορική και θρησκευτική σημασία. Ο Ιορδάνης έχει σχέση και με την διεθνή ασφάλεια. Νομίζω λοιπόν ότι η συζήτηση αυτή ε, θα πρέπει να οδηγήσει στην ε, διάσωση του ποταμού και ε, για να γίνει κάτι τέτοιο δεν πρέπει να καταδικάζουμε τη μία ή την άλλη πλευρά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το άρθρο ε του ψηφίσματος δεν είναι σε άμεση σχέση με το θέμα και θα οδηγήσει σε δυσάρεστες συνέπειες η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές συνέπειες, να οδηγήσει ακόμα και στην πλήρη καταστροφή του ποταμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με τις ειρνευτικές διαπραγματεύσεις. Κυρία Ντεκάιζερ. Θέλετε να συμμετάσχετε στη διαδικασία Κατστιάη. Uh, Mr. Melcher. Πρόεδρε, γνωρίζουμε ότι ο Ιορδάνης ε, έχει μεγάλη σημασία για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ε, ο Ιορδάνης μπορεί πράγματι και συνέβαλε κατά το παρελθόν στην ειρήνη. Στη Συρία όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν φόβοι. Ισραήλ, ε, το Ισραήλ θα μπορούσε να αφαιρέσει, να αποσπάσει από την Συρία τα ύδατα και γι' αυτό το Ισραήλ δεν επιστρέφει τα έψαμα του Κολάν στην Συρία. Εάν λοιπόν τελικά θεωρήσουμε ότι ο Ορδάνη αντί για ποταμό ε, έχει καταλήξει να είναι αυλάκι, όπω σα είπα, ε, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δεχθούμε και ε, ότι η περιοχή εκεί είναι έρημο. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα επιδεινωθεί τα μάλα. Η Χαμά είναι εκείνη η οποία ε, μιλάει ε, κυρίως για το θέμα του Ιορδάνη αλλά η λειψιδρία αφορά και άλλους ε, που ενδιαφέρονται για την περιοχή γιατί το δυναμικό αυτό της σύγκρουσης είναι όλο και πιο έντονο και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στη στρατηγική μας. Δύο, τελευταία γορτές, ο κυρία Κάιζερ και κυρία Μεντέτσεβα. Κυρία Κάιζερ, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που με αφήνετε να διευκρινίσω κάτι το οποίο δεν είχα την ευκαιρία να διευκρινίσω προηγουμένω. Δεν ήμουν ίσω αρκετά πιστική. Το θέμα τη εκμετάλλευση, τη υπερεκμετάλλευση από του επίκου του Ισραήλ. Να θυμίσω την ειδική έκθεση που εγκρίθηκε και από τη συνέλευση Euromed για την κατάσταση των υδάτων στη Μέση Ανατολή και η οποία παραθέτει στην έκθεση της Παγκόσμιας τράπεζας, περιορισμός στην πρόσβαση των Παλαιστινίων και της ε, διεθνούς αμνηστίας για το θέμα του νερού στην ίδια περιοχή. Μιλά, μιλούν οι τρεις ε, εκθέσεις για την υπερεκμετάλλευση κατά τρεις-τέσσερις φορές παραπάνω από τους Ισραηλινούς επίκους. Αυτό λοιπόν που ανέφερα δεν είναι δικό μου σχόλιο, είναι απολύτως τεκμηριωμένο, δεν είναι προσωπική άποψη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας υπεύθυνο εταίρος. Αναλαμβάνει τις ευθύνες της στα πλαίσια της εξωτερικής της πολιτικής. Είναι δωρητής για προγράμματα και σχέδια στη Μέση Ανατολή. Συμμετέχει επίσης στην ειρηνευτική διαδικασία εκεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εκπονήσει μια στρατηγική για τον Ιορδάνη ποταμό που τόσο μεγάλη σημασία έχει για την περιοχή. Οι φίλοι της γης, η οργάνωση αυτή, πριν από ένα μήνα προειδοποίησαν για το ότι θα σταματήσει να έχει νερό η Ορδάνης μέσα σε ένα χρόνο. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικέ συνέπειες θα έχει αυτό για την περιοχή και πόσο μεγάλη απειλή είναι για τι ζωέ των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί. Πέρα λοιπόν από τα γεγονότα, και ω σύμβολο ο Ιορδάνη ποταμό είναι πολύ σημαντικός. Είναι σύμβολο για τις αξίες μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και εμείς να δείξουμε ότι έχουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση σε προβλήματα όπω αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη. Όλοι ζητούν να καταβληθούν κοινέ προσπάθειε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ σωστά εφιστά την προσοχή ε, στο ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ε, προσέγγιση συνεργασία σε αυτή την περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προάγει το πνεύμα συνεργασία ε, με το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υδάτινων πόρων στην Μέση Ανατολή. Το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί στη πηγή, στη ρίζα και όχι μόνο στις εκβολές του ποταμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί η λειψιδρία στην περιοχή και ε, για να διαφυλαχθεί, να προστατευτεί το περιβάλλον, να διαφυλαχθεί το πόσιμο νερό για τους ε, κατοίκους της ε, περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει δραστηριότητες που συμβάλλουν, θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση του Ιορδάνη στο μέλλον και επίσης ε, σε μια κοινή διαχείριση της ε, λεκάνης απορροής του ποταμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει το διάλογο, να προάγει την διασυνοριακή συνεργασία σε θέματα υδάτων ανάμεσα στους ε, διάφορους ε, γείτονες ε, της περιοχής, συμβάλλοντας την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Είναι λοιπόν σημαντικό και οι ίδιες οι όμορες χώρες να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να επιφέρουν μια ισορροπία ανάμεσα στους πόρους και τη ζήτηση. Αυτό δεν αφορά μόνο τις κυβερνήσεις, αλλά και την κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη έχουμε μεμονωμένες επιχειρήσεις αλλά και κοινότητες που καλούνται να συμβάλλουν ε, στην βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πρόκληση για όλους μας. Προτάσεις ψηφίσματος για την περάτωση αυτής της συζήτησης. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. Διακόπτουμε. We'll suspend the, uh, the session until 6 o'clock for just for a few minutes